Ευχαριστώ. Με ενημέρωσαν οι αρμόδιες τσεχικές αρχές ε, για την εκλογή του κ. Βόησεκ Βίλερ που θα, θα αντικαταστήσει τον κύριο Γίζη Χάβελ, τον αποβιώσαντα, από την 9η Ιουλίου. Με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 θα γίνει η... Ε, ε, ο έλεγχος των ασυλιών και των διαπιστευτηρίων για να επιβεβαιωθεί η εντολή του. Θα προσπαθήσω να μιλάω πιο κοντά στο μικρόφωνο για τα πρακτικά. Εφόσον έχει υπογράψει τη δήλωση ότι δεν έχει άλλη σύμβατη με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή θέση, θα αναλάβει ο κύριος Βάζεχ Μίναρτ τα καθήκοντά του μαζί με τα προνόμια και τις ασυλίες που συνοδεύουν την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. έχω λάβει από τον κύριο Βίκτορ Σπάτσιτς ε, μία αίτηση για την πράσπιση της ε, ε, βουλευτικής του ασυλίας με βάση το άρθρο 6.2 θα παραπευθεί στην αρμόδια νομική επιτροπή που είναι η νομική επιτροπή. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες μου έδωσαν τον κατάλογο για τους διορισμούς στις διάφορες επιτροπές. Θα δημοσιευθούν στα πρακτικά και αν δεν διατυπωθούν ενστάσεις μέχρι την έγκριση στο πρακτικό θα θεωρώ